Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Αγαπητή κυρία Μπλινκεβιτσιούτε, καλώς ήρθατε στην ακρόαση αυτή που αποτελεί μια ευκαιρία για τα μέλη τόσο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ όσο και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα της Γυναίκας να ακούσουν τους προσκεκλημένους μας εμπειρογνώμονες όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας του 2012-29 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει ελάχιστες προδιαγραφές για τα δικαιώματα, τη στήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών. Έτσι ανταποκρινόμαστε στην ε, ανάγκη για προστασία και στήριξη των Ευρωπαίων πολιτών που επειδή ταξιδεύουν, ζουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό μπορεί να καταλήξουν θύματα εγκληματικών ενεργειών σε μια διαφορετική χώρα από τη δικιά τους. Η οδηγία αυτή λοιπόν διασφαλίζει ότι τα άτομα που έχουν καταστεί θύματα τέτοιων εγκληματικών ενεργειών θα μπορούν να προστατεύονται κατάλληλα και θα τυχαίνουν της κατάλληλης αρρωγής στην άλλη χώρα που βρίσκονται. Οι χώρες μέλη έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις της οδηγίας, έπρεπε να το κάνουν έτσι κι αλλιώς μέχρι τις 16 Νοεμβρίου του 2015 και έχουν ενσωματώσει την οδηγία αυτή. Στην ακρόαση αυτή θα ακούσουμε τι μέτρα έχουν πάρει τα κράτη-μέλη για να επιτρέψουν στα θύματα να τύχουν αναγνώριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων υπό την οδηγία αυτή και πώς λειτουργούν τα πράγματα σε εθνικό επίπεδο, πώς έχει προχωρήσει η εφαρμογή, με τι δυσκολίες κτλ. Έτσι θα δούμε τι αλλαγές μπορεί να χρειάζονται ή τι πρέπει να προσθεθεί. Η, η, ακρόαση αυτή θα βοηθήσει να εκπονήσουμε και την επόμενη έκθεσή μας που θα συνταχθεί βάσει του άρθρου 55 από τους συνεισηγητές των δύο αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Θα δώσω το λόγο στην συνπρόεδρό μου, την κυρία Μπλίνκεβιτσιούτη. Και επαναλαμβάνω ότι χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Η κυρία Μπλίνκεβιτσιούτη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στάνισεφ και καλωσορίζω εδώ τα μέλη και των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών. Η οδηγία έχει ως στόχο να προστατεύει όλα τα θύματα εγκληματικών ενεργειών, αλλά έχει και μία διάσταση που αφορά το γένος, δηλαδή αφορά και την βία σε βάρος των γυναικών, την ε, φιλική βία στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ένα από τα στοιχεία κλειδί της οδηγίας είναι ότι βάζει τα θύματα στο κέντρο κάθε εγκληματικής ε, δικαστικής διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο μάρτυρες σε αυτή τη διαδικασία, αλλά πρέπει να τυχαίνουν στήριξη και βοήθειες καθ' όλη την δικαστική διαδικασία. Και είναι ζωτική σημασία σε αυτό όταν μιλάμε για θύματα βίας σε βάρος των γυναικών ή για ενδοοικογενειακή βία. Από την άλλη, δεν πρέπει οι γυναίκες και τα παιδιά να γίνονται για δεύτερη φορά θύματα κατά τη διάρκεια των ε, δικαστικών διαδικασιών, ε, επειδή είναι θύματα εγκληματικών ενεργειών. Και οι γυναίκες ε, και τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματα που έχουν και για την κατάσταση όσον αφορά τον θήτη. Η εφαρμογή από τα κράτη-μέλη των δικαιωμάτων αυτών που αναφέρονται στην οδηγία αποτελούν και τον, το αντικείμενο του σχέδιου έκθεσης που ετοιμάζουν οι δύο συνεισηγητές. Είμαι σίγουρη ότι η ακρόση αυτή θα μας βοηθήσει να συλλέξουμε πληροφορίες για το έργο μας. Θα περάσουμε στο πρώτο πάνελ. Πρόκειται για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες στην εφαρμογή της οδηγίας αυτής που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Θα ακούσουμε παρουσιάσεις της, ε, όσον αφορά την οδηγία αυτή. Υπάρχει μελέτη που έχει ετοιμάσει μια ομάδα ερευνητών ε, από το Κέντρο Στρατηγικής και Αξιολόγησης Υπηρεσιών ενώ την αρχική ανάλυση την έχει ετοιμάσει το δικό μας το EPRS. Θα δώσω το λόγο επίσης και στους ερευνητές του Κέντρου Στρατηγικής. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Στέφαν Κράτσερ και την Εζενή Λαλεντεμός. Και οι δύο επιτροπές ασχοληθήκαμε με την προετοιμασία της αξιολόγησης της εφαρμογής που ετοίμασε το PRS και θα μας παρουσιάσει τα πορίσματα. Η κυρία Εζενή Λάλ Ντεμός πρώτα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ξεκινάει ο μιλητής. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη στήριξη των θυμάτων ανά την Ευρώπη. Ξεκίνησε ο κύριος Κρέτσερ και όχι η κυρία Λάλντεμος. Να, η μελέτη μας. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν την ε, οδηγία, θα σας πω ποια είναι τα στοιχεία κλειδί στην έρευνά μας, τα πορίσματά μας. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο, την Εζενή, η οποία θα σας παρουσιάσουν τα πορίσματά μας για οριζόντια ζητήματα, όπως είναι η ατομική αξιολόγηση που είναι υποχρεωτική τώρα από την οδηγία και θα αναφερθώ και σε μερικά ειδικά θέματα που έχουν να κάνουν με εγκλήματα όπως είναι η τρομοκρατία. Τέλος θα παρουσιάσουμε τα συμπεράσματά μας και τις συστάσεις μας. Συνολικά πιστεύουμε ότι η οδηγία ήδη έχει θετικό αντίκτυπο σε πολλές χώρες μέλη. Όμως υπάρχει διαφοροποίηση. Και θα εξηγήσουμε αργότερα τι είναι αυτό το οποίο επηρεάζει και οδηγεί σε αυτές τις διαφορές. Και μετά θα σας μιλήσουμε για τις συστάσεις μας όσον αφορά τη μελλοντική εφαρμογή της οδηγίας. Λοιπόν, όσον αφορά την ε, μελέτη πεδίο εφαρμογής, ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλευτικό Κέντρο Ερευνών και αναφέρεται στην εφαρμογή της οδηγίας η οποία καθορίζει ελάχιστε προδιαγραφέ στα δικαιώματα τη στήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών. Η αξιολόγηση λοιπόν που κάναμε ε, αξιολόγησε την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία στις 27 χώρες ε, μέλη που έπρεπε να ενσωματώσουν την οδηγία. Η Δανία δεν οφείλει να το κάνει αυτό γιατί έχει ένα opt-out, εξαιρείται. Και έπειτα κοιτάξαμε και στην πράξη επιτόπου πώς έγινε η ενσωμάτωση αυτή σε 12 χώρες μέλη δειγματοληπτικά. Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια ποικιλία χωρών, τόσο γεωγραφικά όσο και βάση κουλτούρας που έχει Βέλγιο, Τσεχία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Ισπανία και Σουηδία. Μετά προσπαθήσαμε να εκτιμήσουμε κατά πόσο υπάρχει συνοχή, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και προσθέμενη αξία τώρα που ενσωματώθηκε η οδηγία. Η έρευνα έγινε Ιούνιο με Δεκέμβριο του 2017 και συνδυάστηκε με συνεντεύξεις, με online έρευνες και επαφές με διάφορες ομάδες. Η οδηγία λοιπόν αντικαθιστά προηγούμενες αποφάσεις πλαίσιο του 2001 και έχει σαν στόχο να ενισχύσει τα δικαιώματα των θυμάτων ανεξάρτητα με το που έλαβε χώρα το έγκλημα και ανεξάρτητα από την υπηκότητά τους ή τον χώρο διαμονής τους. Η οδηγία επίσης δίνει έναν ευρύ ορισμό στον όρο θύμα. Είναι οποιοδήποτε ο οποίος έχει πληγεί είτε φυσικά, είτε πνευματικά, είτε οικονομικά και περιλαμβάνει και τα μέλη της οικογένειας στην περίπτωση που υπάρχει θάνατος κατόπιν της εγκληματικής ενέργειας. Η οδηγία έπρεπε να ενσωματωθεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2015 στις χώρες μέλη. Στην πράξη τους τελευταίους έξι μήνες ενσωμάτωσαν την οδηγία πολλές χώρες. Οπότε καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στην πράξη. Ζητήθηκε πάντως από τις χώρες μέλη να πούνε τι αλλαγές έχουν γίνει στις υπηρεσίες τους και έπρεπε να στείλουν τις απαντήσεις τους μέχρι τον Νοέμβριο του 2017. Λοιπόν, Ποια είναι τα κύρια πορίσματα. Όπως είπα και πριν, οι περισσότερες χώρες έχουν ήδη ενσωματώσει την οδηγία στην εθνική του νομοθεσία με μερικές μόνο εξαιρέσει. Ιρλανδία, Σλοβενία, για παράδειγμα, φέτο θα γίνει αυτό. Οι χώρες που δεν έχουν ενσωματώσει την ε, οδηγία το έχουν κάνει εξαιτία εσωτερικών ε, περιπλοκών ε, που αφορούν αυτές τις χώρες και μόνο. Αν δούμε τώρα πώς στην πράξη εφαρμόζεται η οδηγία, έχουμε καταλήξει σε τρεις κατηγορίες χωρών. Υπάρχουν οι χώρες εκείνες όπου πριν την οδηγία δεν είχαν αρκετά ανεπτυγμένο σύστημα στήριξης των θυμάτων. Τσεχία, Λιθουανία και μια άλλη κατηγορία. Μάλλον σε, αυτές τις, σε αυτή την κατηγορία ε, βέβαια υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις. Έπειτα υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν ε, ξόδεψαν περισσότερα χρήματα για να εφαρμόσουν την οδηγία Ισπανία, για παράδειγμα. Οπότε οι επιπτώσεις τη οδηγίες είναι ελάχιστες. Και υπάρχουν ε, και οι χώρες που είχαν ήδη ένα καλά αναπτυγμένο σύστημα προστασίας των θυμάτων και πριν την οδηγία, η Αυστρία ή η Σουηδία, και εκεί οι επιπτώσεις δεν ήταν τόσο αισθητέ. Δεν ε, αυξήθηκε τόσο πολύ το επίπεδο προστασίας, απλώς διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της προστασίας αυτής. Τώρα θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο την Ευζενή. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Η μελέτη μας κατέληξε ότι μία από τις καινοτομίες της οδηγίας αυτής είναι η διάθεση μεταφραστών και διερμηνέων. Και φαίνεται ότι πρόκειται για ένα τεράστιο επίτευγμα διότι αντιμετωπίζεται έτσι και η πολυπλοκότητα των διασυνοριακών εγκλημάτων, αλλά αντιμετωπίζεται έτσι και το ίδιο το νόημα της οδηγίας που ήταν έχουν τα ίδια δικαιώματα όλοι οι πολίτες θύματα εγκλημάτων ανεξάρτητα από το που έλαβε χώρα το έγκλημα. Μια άλλη καινοτομία είναι εκείνη της ατομικής αξιολόγησης. Στη πράξη διαφέρει βέβαια η κατάσταση από τη μία χώρα στην άλλη. Παρ' όλα αυτά διαπιστώσαμε ότι περισσότερε χώρε μέλη έκαναν προσπάθειες να επεκτείνουν τις ατομικές αυτές αξιολογήσει σε παντό είδου εγκλήματα και θύματα. Υπάρχουν και δύο διαφορετικές προσεγγίσεις από τις χώρε μέλη για να στηρίξουν τα θύματα. Η πρώτη είναι το σενάριο opt-out. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι χώρες μέλη προσφέρουν έτσι και αλλιώς προστασία στα θύματα το Βέλγιο και η Γαλλία ακολουθούν αυτό το σύστημα. Από την άλλη μεριά υπάρχει η προσέγγιση opt-in, που σημαίνει ότι τα θύματα δεν παίρνουν αυτόματα προστασία, αλλά θα πρέπει να ζητήσουν την προστασία αυτή. Αυτό ισχύει σε χώρες μέλη όπου ε, το σύστημα προστασίας των θυμάτων είναι λιγότερο ανεπτυγμένο. Τέλος, η οδηγία ε, υπογραμμίζει και διαδικαστικά δικαιώματα όπως είναι εκείνο της αποζημίωσης για θύματα εγκλημάτων που εμπίπτουν στα, στα πλαίσια της δικαστικής διαδικασίας. Τώρα, ποιες είναι οι δυσκολίες στην πράξη. Εξακολουθεί να, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια κενά και κάποιες αδυναμίες στο σύστημα προστασίας των θυμάτων. Η αστυνομία, για παράδειγμα, πολλές φορές δεν στέλνει τα θύματα στις οργανώσεις στήριξη των θυμάτων, που σημαίνει ότι τα θύματα δεν παίρνουν τελικά τη βοήθεια από το σύστημα το οποίο δικαιούνται. Και στο τέλος, έτσι γίνεται λιγότερο αποτελεσματική η οδηγία. Πρέπει να υπάρχει η διαθεσιμότητα αυτή και η πρόσβαση των θυμάτων στο σύστημα, αλλά δυστυχώ δεν γίνεται αυτό σε όλε τι χώρε. Δεν καταφέρουν πάντα να ασκήσουν τα δικαιώματά του, περισσότερε φορέ γιατί δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά του ή γιατί δεν γνωρίζουν τι υπηρεσίε υπάρχουν για να ε, τα στηρίξουν. Και τέλο διαπιστώσαμε ότι η εκπαίδευση, κατάρτιση των ε, αρχών ε, των υπηρεσιών που ασχολούνται με αυτό το θέμα είναι κάτι ζωτική σημασία. Αλλά δυστυχώ δεν συμβαίνει παντού. Δεν είναι διαθέσιμη τέτοια κατάρτιση σε όλε τι χώρε για του αρμόδιου. Τώρα στη μελέτη μας εξετάσαμε και ειδικέ ε, περιπτώσεις. Η πρώτη ήταν τα θύματα της τρομοκρατίας. Εδώ υπάρχει πολύ το διασυνοριακό θέμα. Στην Βαρκελόνη, για παράδειγμα, είχαμε 30 διαφορετικές υπηκότητες θύματα της πρόσφατης τρομοκρατικής επίθεσης. Τα θύματα της τρομοκρατίας συνήθως δεν έχουν ένα ειδικό σύστημα προστασίας. Μετά τις τελευταίες τρομοκρατικές ενέργειες όμως στην Ευρώπη άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα και οι χώρες μέλη έχουν προσαρμόσει τα εθνικά τους πλαίσια για να αντιμετωπίσουν και τις ανάγκες των θυμάτων αυτών. Στη Γαλλία και το Βέλγιο κυρίως προθήθηκαν τέτοια συστήματα και προσαρμόστηκαν. Όσον αφορά τώρα τη βία που έχει να κάνει με το φύλλο, υπάρχει καλή προστασία, διαπιστώσαμε, αν και εξακολουθούν οι περιπτώσεις αυτές να μην φτάνουν στις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που δεν καταγγέλλονται. Επίσης ότι δεν υπάρχει αρκετή προστασία στα θύματα της ορτορικής μίσους. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι η οδηγία έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές και καινοτομίες, αλλά διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Επίσης είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι πολλές χώρες μέλη εξακολουθούν να βασίζονται στον εθελοντισμό για να προσφέρουν τέτοιου είδου υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι συχνά δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς ή δεν έχουν αρκετό προσωπικό αυτές οι υπηρεσίες από συστάσεις έχουμε να πούμε ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση στα θύματα και για τα δικαιώματά τους, αλλά και για τις διάφορες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τα θύματα πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους όταν βρίσκονται και στο εξωτερικό. Γι' αυτό προτείνουμε να υπάρχει καλύτερη σήμανση. Είναι κάτι το οποίο ισχύει στην Ουγγαρία. Επίσης, η οικοδόμηση ικανοτήτων και η κατάρτιση είναι σημαντικά ζητήματα και να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τις καταγγελίες τέτοιων εγκλημάτων. Και για να ολοκληρώσω θέλω να πω ότι οι χώρες μέλη θα έπρεπε να επικεντρωθούν να ενθαρρύνουν την ίδια, την εξίσου σημαντική αντιμετώπιση όλων των ειδών εγκλημάτων. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω και με το εξής διαπιστώσαμε ότι η οδηγία δείχνει θετικό αντίκτυπο στις περισσότερες χώρες ε, μέλη. Βέβαια σε κάποιες ενσωμάτωση έχει γίνει πολύ αργά, οπότε μας χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε παρετέρω την κατάσταση. Οπότε αξίζει τον κόπο σε λίγα χρόνια να ξανακάνουμε την ίδια αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σινή και κύριε Στέφαν Κράουτσερ για την παρουσίασή σας. Και τώρα να δώσω το λόγο στους συνεισηγητές. Τερέζα Χιμένες Μπεσερίλ Μπάριο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ παίρνει το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλους τους παρόντες στην ακρόαση αυτή που είναι τόσο σημαντική για τα δικαιώματα, την προστασία και τη στήριξη των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών. Ακούσαμε ότι τα θύματα διαφέρουν μεταξύ τους πολύ, όπως επίσης και τα εγκλήματα. Έχουμε εδώ μαζί μας τη συντονίστρια μια γυναίκα που έχει αγωνιστεί πάρα πολύ όσον αφορά την καταπολέμηση της λαθροδιακίνησης και της ε, λαθροεμπορίας. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ μετά από τις επιθέσεις της Βρυξέλλες. Έχουμε και θύματα εδώ από την Ουγγαρία και άλλα από την Ισπανία, από τη χώρα των Βάσκων, για να να μας μιλήσει για την εμπειρία της. Και θέλω να ευχαριστήσω και τη συνεισηγήτρια βεβαίως με την οποία συνεργαστήκαμε πολύ αρμονικά. Ευχαριστώ και την Υπηρεσία Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το EPRS, για την έκθεσή του και το πώς οι χώρες μέλη έχουν εφαρμόσει μέχρι τώρα την οδηγία αυτή. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έχει παρουσιάσει ακόμα τη δική της έκθεση για αυτήν την εφαρμογή, η έκθεση του EPRS είναι πολύ χρήσιμη για μας. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζω να μας εξηγήσει πότε θα έχουμε τη δικιά της την έκθεση. Από τότε που έφτασα στο Κοινοβούλιο και είδα ότι δεν υπάρχει νομοθεσία για τα θύματα, μόνο μία απόφαση πλαίσιο που ουσιαστικά δεν εφαρμόζονταν, ήρθα σε επαφή με την Επίτροπο Ρέντινγκ τότε για να ετοιμάσουμε αυτό το πακέτο για τα θύματα. Οποιοςδήποτε μπορεί να γίνει θύμα Έχουμε 75 εκατομμύρια θύματα, είτε πρόκειται για μικρά εγκλήματα, είτε πρόκειται για θύματα οργανωμένου εγκλήματος, τρομοκρατίας κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να βοηθήσουμε τα θύματα. Ήμουν εισηγήτρια στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και θυμάμαι τι εγώ να δώσαμε τότε στις διαπραγματεύσεις, στους τριμερείς διαλόγους για τα δικαιώματα των θυμάτων. Καταφέραμε να συμπεριλάβουμε κάτι πολύ βασικό, όπως είπε και ο Πρόεδρος, τι ελάχιστε προδιαγραφέ, που είναι και ο τίτλο τη οδηγία. Οι ελάχιστε προδιαγραφέ είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν όμω. Γιατί πρέπει ο άλλο να σε καταλάβει όταν είσαι θύμα τέτοια εγκληματική ε, ενέργειας, να καταλάβει τι λες και να μπορέσεις να φτάσεις στην πρώτη βασική υπηρεσία αρχή που μπορεί να σε προστατεύσει. Χρειάζεται απλή γλώσσα. Είχαμε τις πρώτες αρχές ε, με μια υπηρεσία για το τι πρέπει να λένε τα θύματα, γιατί ένα θύμα όταν φτάνει σε μια τέτοια υπηρεσία καλά καλά δεν γνωρίζει που βρίσκεται. Οπότε πρέπει να καταλάβει τι επιπτώσεις έχει επαφή αυτή για το μέλλον. Και πρέπει επίσης να μπορεί κάποιος να καταγγέλει και να παίρνει αντίγραφο της καταγγελίας. Σε μερικές χώρες δεν την παίρνει. Απλώς αναφέρεται η καταγγελία σε ένα μητρό και δεν υπάρχει τίποτα για το θύμα. Έπειτα, η διερμηνία και η μετάφραση. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να έχει στη γλώσσα του πληροφορίες για τη δικαστική διαδικασία. Ένας πολύ σημαντικός τομέας που ξεκολουθεί να είναι ζωτική σημασία είναι αυτό που ονομάσαμε τότε ατομική αξιολόγηση που είναι ζωτική σημασία προκειμένου να καταλάβουμε ποιε είναι οι δικέ ανάγκε του κάθε θύματο. Έχουν γίνει πρόοδοι στις διάφορες χώρες μέλη, διοικητικά και νομοθετικά όσον αφορά την ατομική αξιολόγηση. Όμως ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η ατομική αξιολόγηση, όπως μας είπαν και οι συνάδελφοι εδώ, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ακόμα και στην ίδια χώρα διαφέρει από τη μία πόλη στην άλλη, από τη μία περιφέρεια στην άλλη. Οπότε τελικά το θύμα δεν έχει την ίδια στήριξη παντού. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Κάτι άλλο είναι ότι οι χώρες δεν δέχονται να αναλάβουν την ευθύνη για τα θύματα τρομοκρατίας, π.χ. η χώρα, δεν δέχεται ότι τελικά αυτή είναι υπεύθυνη για τη ζημιά που έχει πάθει το θύμα. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό και θα επιμείνουμε σε αυτό και το βάζουμε στην έκθεση, είναι οι εκστρατείες ενημέρωσης και συνειδητοποίησης awareness raising campaign που συνοδεύουν την εφαρμογή της οδηγίας. Δεν υπάρχει ενημέρωση σε μια απλή γλώσσα που να μπορεί να καταλάβει το θύμα. Γιατί δεν πάνε τα θύματα, δεν πάνε γιατί δεν καταλαβαίνουν, δεν υπάρχει εκστρατεία στα περιοδικά, στις εφημερίδες, στην τηλεόραση τα θύματα δεν γνωρίζουν ότι έχουν τέτοια δικαιώματα να πάνε να καταγγείλουν και να ζητήσουν στήριξη. Έπειτα χρειάζεται και οικονομική στήριξη και δεν υπάρχει αρκετό συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών ε, των δικαστικών, των αστυνομικών, ε, εισαγγελία κλπ. Μερικέ φορέ κάτι ξέρει η αστυνομία που δεν το ξέρει όμω ο δικαστή, οπότε σπάει η αλυσίδα. Και υπάρχει και έλλειψη κατάρτισης για τους επαγγελματίες του κλάδου. Σωστά, με την ε, συνεισηγήτρια την κυρία Μίλνερ πιστεύουμε ότι πρέπει να υπογραμμιστεί στην έκθεση η εφαρμογή της οδηγίας με τα σφάλματα τα οποία γίνονται μέχρι τώρα που πρέπει να σταματήσουν. Θα έλεγα λοιπόν για να ολοκληρώσω ότι θα πρόσθετα ειδικέ συστάσεις για τα δικαιώματα των θυμάτων τρομοκρατίας. Μετά τα τελευταία ακούσαμε λίγα γίνανε γιατί δεν υπήρχε εμπειρία. Δυστυχώς η χώρα μου ναι έχει εμπειρία εδώ και χρόνια. Και εγώ είμαι θύμα τρομοκρατίας όταν το 98 δολοφόνησε τον αδερφό μου και την γυναίκα του Ιέτα και άφησε ένα παιδί ορφανό. Ήταν πολιτικός, αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Να εδώ συνάδελφος που είχε ε, στρατιώτη πατέρα είναι θέμα και το άλλο θέμα θέλω να πω, το άλλο θύμα θέλω να πω ότι οποιοδήποτε μπορεί να καταστεί θύμα της τρομοκρατίας και στην Ευρώπη δυστυχώς δεν έχουμε δώσει αρκετή σημασία στα θέματα δεν δώσαμε εγγυήσει για τα δικαιώματά τους στο Βέλγιο έγινε μια ακρόαση για τα θύματα του 2016 και είπαν ότι δεν πήραν ούτε οικονομική ούτε ψυχολογική στήριξη ένιωσαν εγκαταλελειμμένοι. Και είναι τρομερό αυτό. Γιατί υπήρχε ήδη οδηγία για τα θύματα και οι χώρε μέλη ήξεραν ότι έπρεπε να την εφαρμόσουν και έπρεπε να το έχουν κάνει και δεν το έκαναν. Και δεν δέχονται και την ευθύνη τους. Όλα τα ζητάνε από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ναι, αλλά στο αεροδρόμιο όπως έγινε εδώ ή αλλού μπορεί να έχεις ασφάλεια ιδιωτική κτλ. Αλλά δεν είναι θέμα της ασφαλιστικής εταιρείας. Η επίθεση έγινε κατά της δημοκρατίας, κατά των αξιών που στηρίζουμε και κατά της χώρας μέλους. Και τελικά ο τελευταίος υπεύθυνο είναι η χώρα μέλη που μέλος που πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Για να αποφύγουμε λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις που είναι προστάτευτο το θύμα τρομοκρατίας, όπως μας λένε πολλοί, οι χώρες πρέπει να φροντίσουν για κατάρτιση στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναλάβει να βοηθούν τα θύματα τρομοκρατίας και πρέπει να υπάρχει κάποιος υπεύθυνο και όχι να στέλνουν το θύμα από τη μια μέρα στην άλλη, τη μια στο γιατρό, τον ένα, την άλλη στον άλλο, την άλλη στον τρίτο και τελικά να νιώθουν ξανά και ξανά θύματα κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε η ιατρική και ψυχολογική βοήθεια για να ξεπερνάει κανείς το τραύμα. Αποτελεσματικά όμως, όχι γραφειοκρατικά για να μπορεί κανείς να συμπληρώσει ένα χαρτί. Ζητούμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες αποκατάσταση ώστε ό,τι ζημιά έχει υποστεί το θύμα να μπορεί να την ξεπεράσει, να μπορεί να ξαναβρει δουλειά, οτιδήποτε χρειάζεται. Χρειάζεται επίσης και μια τηλεφωνική γραμμή η οποία να Πείτε αμέσως έτσι και υπάρξει τρομοκρατική επίθεση και να υπάρχει βοήθεια σε πολλέ γλώσσε. Γιατί όπω είπαμε στι τρομοκρατικέ ενέργειε, όπω έγινε και στη Βαρκελόνη, είχαμε διαφορετικέ ε, υπηκότητε, 30 διαφορετικέ των θυμάτων. Να ενημερώνονται τα, ε, οι συγγενεί. Εμένα ήρθαν σε επαφή ε, άνθρωποι που μου είπαν ότι δεν ξέρανε πού είναι το παιδί του, γιατί ήταν από άλλη χώρα. Έχουμε εδώ δύο θύματα, όπως σας είπα και πριν, της τρομοκρατίας, που θα μας πούνε και αυτοί τι πιστεύουν ότι είναι το πιο χρήσιμο. Και έχουμε και άλλους που θα μας μιλήσουν για άλλου είδους ε, εγκληματικές ενέργειες, θύματα των οποίων είναι. Μας μένει πολλής δρόμος για να πετύχουμε τη μνήμη, την αλήθεια, την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη για όλα τα θύματα. Πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας όλοι για να προσφέρουμε τη στήριξη αυτή που όλοι αξίζουν. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χιμένες Μπεσερίλ Μπαριό, εισηγήτρια της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Τώρα, η κυρία Αγγέλικα Νίπλερ από την Επιτροπή Γυναικών. Ευχαριστώ τους φιλοξενούμενους για τη διοργάνωση αυτής της ε, εκδήλωσης, λέει η κυρία Μίλνερ. Θα συνεχίσω από εκεί που η κυρία Μπαριό σταμάτησε. Ε, κάνε μια πολύ καλή επισκόπηση περισσότερο τη γυναικεία πλευρά καλύπτει αυτό το κομμάτι της έκθεσης. Θα ήθελα να καλύψω εγώ τη γυναικεία πτυχή. Κάτι γενικό. Είμαι νομικός εγώ και θα πρέπει γενικά να αποδεχθούμε την αλήθεια. Η κοινωνία εστιάζεται επί εκείνου που διαπράττει το αδίκημα, το αγκλήμα. Εστιαζόμεθα επί, εκείνου, επί του δράστου και προσπαθούμε το να επανατάξουμε στην κοινωνία. Λυσμονούμε όμως τι γίνεται με το θύμα αυτό είναι κάτι που η ποινική νομοθεσία όλων των κρατών ε, δεν το προσέχει επαρκώς. Είναι και η ώρα να αρχίσουμε συζήτηση όσον αφορά και το θέμα αυτό, το θύμα. Αναφέρατε στη σύντομη παρουσίασή σας κάτι σημαντικότατο, ότι δεν καταγγέλλεται επαρκώς οικιακή βία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα κοινό για όλες τις κοινωνίες και όλα τα κάτι μέλη. Η οικιακή βία, η ενδιοοικογενειακή βία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αντιμετωπίζεται, αλλά δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα. Το εμπόριο ανθρώπων, ε, κυρίως βασικά θύματα είναι γυναίκες αυτού. Και έχω μια ερώτηση. Κάτι που έχει αναφερθεί στα μέσα ενημέρωσης δεν έχει συζητηθεί στο Κοινοβούλιο Ετοιμάζουμε απλώς προφορική ερώτηση. Όμως, ενώ δεν έχει ξεκινήσει η συζήτηση, το θέμα είναι το εμπόριο των ανθρώπων και μιλώνω για τους εποχιακούς εργαζόμενους. Που πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως αντιμετωπίζονται στα κράτη-μέλη σαν σκλάβοι. Είναι θύματα, μια ομάδα θυμάτων που δεν έχει φωτιστεί δεν έχουμε ρίξει τον προβολέα πάνω τους. Ετοιμάζεται η προφορική ερώτηση. Ελπίζω να διεξαχθεί στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα συζήτηση. Έχετε κάποια αριθμητικά στοιχεία γι' αυτό. Έχετε εξετάσει αυτό το θέμα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι υπάρχει ισχύουσα νομοθεσία. Οδηγίες. Νομοθετικός πώς λειτουργούν επί χάρτου είναι λογικά τα μέτρα, αλλά δεν εφαρμόζονται. Μπορεί να έχει κανείς την καλύτερη δυνατή νομοθεσία στο χαρτί, άμα δεν εφαρμόζεται όμως δεν βοηθάει. Τα ενδεχόμενα θύματα και τα πραγματικά θύματα. Μπορείτε να το εξετάσετε και αυτό. Είναι πολύ ζήτημα για την ώρα. Και από την πλευρά μου θα προσπαθήσω στην έκθεσή μου να το τονίσω αυτό το πρόβλημα. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μίλναρ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέλαμε να σχολιάσει εν συντομία την εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη-μέλη. Η κυρία Κατερίνα Γιάννησκα, που ηγείται μια ομάδα αρμόδιας για τα δικαιώματα των θυμάτων, στην DG Jost θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να καλωσορίσει την έκθεση του Κοινοβουλίου Πιστεύουμε ότι δίνει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αυτό το σημαντικό εργαλείο στα στο πλαίσιο των δικαιωμάτων ε, των θυμάτων ενσωματώνεται στην Ομοθεσία των μελών και εφαρμόζεται πλήρης και σωστή ενσωμάτωση αυτού του σημαντικού εργαλείου είναι προτεραιότητα για μας, μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κινηθήκαμε τάχιστα τον Ιανουάριο του 2016. Ξεκινήσαμε 16 διαδικασίες επί παραβάση κατά κρατών μελών που δεν κοινοποίησαν εγκαίρως τα εθνικά μέτρα για την ενσωμάτωση οδηγίας. Κάποιες διαδικασίες επί παραβάση δυστυχώς ε, εξακολουθούν. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερα κράτη-μέλη που δεν έχουν ενσωματώσει πλήρως την οδηγία στην ένωμη τάξη τους Πολλή δουλειά γίνεται από την πλευρά μας για να εξασφαλίσουμε την ενσωμάτωση αυτή που πρέπει να είναι πλήρης και ορθή και τέλος να εφαρμόζεται σωστά. Η νομοθεσία είναι ένα τεράστιο μέσο αυτό, πολύ σημαντικό. Αλλάζει όχι μόνο την εθνική ποινική διαδικασία, αλλά απαιτεί τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν και διάφορα συνοδευτικά μέτρα πολλά διοικητικά μέτρα που θα εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή αυτών των διατάξεων στην πράξη. Απαιτεί τα κράτη-μέλη όχι μόνο να ενσωματώσουν συγκεκριμένες διατάξεις στη δική τους ένωμη τάξη, στην ποινική του, στον ποινικό τους κώδικα ή να έχουν συγκεκριμένες πράξεις και διατάξεις για δικαιώματα των θυμάτων, αλλά συχνά απαιτεί και σοβαρή δημοσιονομική υποστήριξη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν πολύ ένα σύστημα στηρίξεως των θυμάτων, σχετικές υπηρεσίες, να διοργανώνεται κατάρτιση για όλα τα άτομα που έρχονται σε επαφή με τα θύματα. Αυτά είναι ένα-δύο παραδείγματα και μόνο. Ένα κομμάτι από τις διαδικασίες επιπαραβάση που συνεχίζονται και γι' αυτό έχουμε αναθέσει εξωτερική μελέτη για να καταλάβουμε το βαθμό των προβλημάτων όσον αφορά την πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας στην ένωμη τάξη και πώς εφαρμόζεται. Παράλληλα, ακολουθούμε και έναν επικοδομητικό διάλογο με τα κρατη Δεν θέλουμε να παραπέμψουμε τα περισσότερα στο δικαστήριο και να έχουμε αποφάσεις κατά αυτών. Θέλουμε τελικά να υπάρχουν διατάξεις που εσωματώνται στην ενόμη τάξη των 100 μελών σωστά και που λειτουργούν στην πράξη. Στον επικοδομητικό διάλογο, λοιπόν, ε, ακολουθούμε διάφορες πρωτοβουλίε με τα κράτη-μέλη. Παραδείγματα. Τέλος του μηνός, 29 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει μια διάσκεψη ψηλού επίπεδου. Θέματα δικαιώματα των θυμάτων. Θα συζητήσουμε ευρέως την εφαρμογή της οδηγίας δικαιώματα των θυμάτων, θα συζητήσουμε το πώς η οδηγία εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Η διάσκεψη ε, θα ξεκινήσει με ομιλία της Επιτρόπου που δείχνει τη σημασία που δίνει στο θέμα αυτό και ότι την υποστηρίζει και η Βουλγαρική Προεδρία θα συμμετάσχει. Ο, Βουλγαρ, ο Βουλγαρος Υπουργός Δικαιοσύνης θα μιλήσει στην αρχή της διάσκεψης. Πέραν από αυτό συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκδικαίων των Θυμάτων. Είναι ένα δίκτυο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το πρόγραμμα JUST. Εκεί συναθρίζονται εθνικοί εμπειρογνώμονες των Υπουργείων Δικαιοσύνης. Στόχος είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Να βοηθήσει κάθε χώρα την άλλη για την εφαρμογή ε, του εργαλείου αυτού που είναι και δύσκολο να εφαρμοστεί. Έχουμε ε, μια πολιτική ενσωμάτωση σε αυτή τη πτυχή σε διάφορε πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Όποτε είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Πώς να επεκτείνουμε Φερρυπίν το μέτρο αυτό και στα θύματα με ειδικέ ανάγκες να υπάρχουν διατάξεις που αντιστοιχούν πλέον επακριβώς τις ειδικέ ανάγκες διαφόρων κατηγοριών θυμάτων όπως θύματα της τρομοκρατίας ένα παράδειγμα είναι αυτό και αποζημιώσεις που δίδονται προστήματα της τρομοκρατίας είναι από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο πρόεδρος, ο κ. Γιούνκερ, πρόσφατα θεώρησε την κυρία Μίρκα σαν ειδική σύμβουλο για τις αποζημιώσεις για τα θύματα των εγκλημάτων. Τα λέω όλα αυτά για να δείτε ότι ασχολούμεθα πάρα πολύ με τα θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων των θυμάτων για τη σωστή ενσωμάτωση στην ενόμη τάξη των κρατών μελών και σωστή υλοποίηση οδηγία. Είναι ύψιστη προτεραιότητα αυτή για μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ με μας μένει πολύς χρόνος. Θα δώσω το λόγο στους κοιόδης συζητητές και στα μέλη. Η κυρία Κοσλόφσκα, Ριέγευ, συγγνώμη, θέλει να πάρει το λόγο. Και παρακαλώ να περιοριστούν σε ένα δίλεπτο τα μέλη της Επιτροπής της ε, παρεμβάσεις τους. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την ακρόαση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω. Θέλω να μιλήσω εκ μέρους της Μαρία Άννα Κοράτσα Μπίλτ, που είναι σκιώδης συγγήτρια εκ μέρους του ΕΛΚ. Και στην αρχή θα ήθελα ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την οδηγία και για όλες τις δραστηριότητε που αφορούν την προστασία των θυμάτων, αλλά επίσης και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Έρευνας του Κοινοβουλίου, την EPRS, για αυτή την πολύ καλή έκθεση που αφορά την εφαρμογή της οδηγίας. Είναι ενδελεχής και επαγγελματική ανάλυση και συγχαρητήρια σε όλες τις χώρες που έχουν σωματώσει την οδηγία στην ενόμη τάξη του. Παρά τις καθυστερήσεις και κάποια προβλήματα, νομίζω ότι στην πράξη τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά. Θα πρέπει να συγχαρούμε και τις ΜΚΟ και όλους τους φορείς και θεσμούς που καθημερινά συνεργάζονται με τα θύματα και που στηρίζουν τα θύματα. Και βέβαια θα ήθελα να προσφέρω την υποστήριξή μας και συνεργασία εκ μέρους της Μαρία Κοράτσα Μπίλτ και όλων των μελών του ΕΛΚ αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τα θύματα, θα το κάνουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και του αγορητέ που ακούστηκαν, την κυρία Χιμένε, την κυρία Εμλίνερ, διότι υπάρχει μια μικρή ομάδα ανθρώπων που ασχολούνται πολύ με το θέμα, είναι πάντα παρόντε στι ακροάσει, πάντα μιλούν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών και για αυτού του ανθρώπου το θέμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Και θα ήθελα να πω ότι αυτή η οδηγία είναι ένα άριστο παράδειγμα κάποιας ενοπίσως και εναρμονίσεως του ποινικού δικαίου στην Ευρώπη. Η κυρία Ρέντινγκ, η Επίτροπος Ρέντινγκ το κατάφερε αυτό και χαίρομαι όλος ιδιαίτερος διότι αυτή η οδηγία δείχνει σαφέστατα ότι η βία κατά των θυμάτων πολύ συχνά είναι η βία κατά των γυναικών. Έχουμε αυτή την έμφυλη διάσταση λοιπόν που είναι σαφέστατη. Επίσης, έχουμε και το νομικό λεξιλόγιο που σχετίζεται με την έμφυλη βία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η δευτερογενής ε, πρόκληση θυμάτων, ε, τα ψυχολογικά προβλήματα των θυμάτων και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία είναι πολύ καλή, δεν είναι τέλεια. Διότι αυτά τα θέματα ε, δημιουργούνται επίσης από την παιδεία, από τα στερεότυπα και εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε κάποιες προσπάθειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, η κυρία Άννα Χέιτ, ε, έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σουηδικά. ειδικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση που κάνατε και τις απόψεις των συναδέλφων. Όπως είπε ε, η συνάδελφος, 65 εκατομμύρια θύματα το χρόνο έχουμε και ανεξαρτήτως είδος εγκλήματος είναι ε, τραγικό για τα ίδια τα θύματα. Οπότε τι να κάνουμε να ταξινομούμε κατά σειρά προτεραιότητας ε, τα θύματα. Δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό. Και θα πρέπει κάτι άλλο να προσφέρουμε μέσα ε, από τη συζήτησή μας. Έχετε πρόβλημα που μιλάω σου ειδικά. 75 million. 75 million. 75 <laughs> εκατομμύρια διορθώνει. Καλά, εγώ είπα 65, 75 ή ακόμη περισσότερο. Επίσης αναφερθήκατε στο εμπόριο στην εμπορία ανθρώπων και που έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία δέκα χρόνια και ε, η τελευταία νομοθεσία χρονολογείται από το 2011 και χάρη σε αυτήν έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερη προστασία. Επίσης έχουμε και στρατηγικές για την εμπορία ανθρώπων για να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη ώστε μεταξύ όλων να ενισχύσουν την προστασία των θυμάτων. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εισηγηθεί καμία στρατηγική ε, για την εμπορία ανθρώπων και έχει εκπνεύσει παλαιότερα το 2016. Τι μήνυμα περνάμε λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον ΟΑΜΗΝ συγείται νέα πολιτική. Περνάει ένα μήνυμα στα κράτη-μέλη αλλά και στου εγκληματίε ότι α, εντάξει δεν είναι και πάρα πολύ σοβαρό, δεν χρειαζόμαστε πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώ ακριβώ, τι προβλέπετε νομοθετικά στα διάφορα κράτη-μέλη. Εσείς κάνατε την πρώτη παρουσίαση, δεν θυμάμαι ακριβώς όπου είστε. Μας μιλήσατε για στατιστικά στοιχεία που έχουν ε, ε, προσαρμοστεί λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου, να δούμε ποια από τα θύματα είναι οι γυναίκες, ποια είναι άντρες. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε και αυτό, γιατί το μεγάλο ποσοστό είναι γυναίκες, κυρίως σε σχέση με την κατοίκο βία και την οικογενειακή βία, δηλαδή και την βορεία ανθρώπων. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να θέλει κάποιο άλλο το λόγο από τα μέλη της Επιτροπής μας. Ε, οι ε, εμπειρογνώμονε θέλουν πολύ σύντομα να απαντήσουν γιατί έχουμε και δεύτερο πάνελ, μην το ξεχνάμε και ε, τρέχει ο χρόνος. Θα απαντήσω και για τους δύο μας στα ερωτήματα των μελών της Επιτροπής. Δυστυχώς όχι. Δηλαδή εμείς ε, ε, δεν ασχοληθήκαμε τόσο πολύ με, την, ε, με το να εκτιμήσουμε τη διάσταση του προβλήματος, αλλά με το πρόβλημα επιτόπου. Έγινε και μία μελέτη για θύματα έμφυλης βίας και τη μεταχείριση είχαν και επίσης για μετανάστες που έπεσαν θύματα δεν ναι, έχει σχέση ε, με εθνικότητα, δηλαδή μέσα στη μελέτη έχουμε και διεπικός τρίτων χωρών. Προκύπτει από τη μελέτη αυτή λοιπόν πως ε, για περιπτώσεις ε, ε, ε πορνείας και οικογενειακής ε, ε, βίας ε, βλέπουμε ότι πρόκειται για δευτερογενή θυματοποίηση, δηλαδή πρώτα εισήλθαν στο εδαφός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει και αυτή η πρόσθετη διάσταση πέρα δηλαδή από αυτή της έμφυλης βίας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντεπρέ θέλει το λόγο. oui, merci, Président. je malheureusement pas participé. Ε, δυστυχώς δεν ήμουν εδώ από την αρχή της συζήτηση. Ε, ήθελα να ε, θέσω μια ερώτηση. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που είχαμε στις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις της Γαλλίας και του Βέλγιου είναι η ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών ανεξαρτήτως προέλευση Στο Βέλγιο, στην τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο και στο μετρό, ήταν 24 διαφορετικές εθνικότητες τα θύματα. Ε, ο μηχανισμός ε, μέχρι στιγμής δεν υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να προσφέρουν ε, ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως ηθαγένειας. τώρα αλλάζει αυτό και το, εσείς μέσα στην πρόταση σας πραγματεύεστε αυτό το ζήτημα, γιατί και πέρα από αυτό έχουμε και άλλα τρία ζητήματα. Αποζημίωση των θυμάτων από το κράτος όπου διεπράχθη η τρομοκρατική ενέργεια. Όταν όμως επιστρέφουν στη χώρα τους δεν υπάρχει εναρμόνιση. Δεύτερον, στη Γαλλία υπάρχει και ταμείο εγγυήσεων. Εγώ είμαι υπέρ ε, ενό ταμείου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να οργανωθούν, όχι να είναι να οργανωθούν καλύτερα οι διαδικασίες αποζημίωσης των θυμάτων. Γιατί πλήττονται οι θεμελιώδες κοινέ μας αξίες, όχι μόνο τα θύματα. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό αλληλεγγύης. Και κάτι άλλο που επίσης είναι σημαντικό και πρέπει να το συζητήσουμε κατά τη γνώμη μου είναι οι διαφορές στα αισθήματα κοινωνικής ασφάλισης και αυτό ε, σχετίζεται με το πρώτο που σας είπα. Κυρία εισηγήτρια, θα κάνετε μια σύνθεση για τη συγκρότηση ε, Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αλληλεγγύης ε, στην εκθεσή σας. Κύριε Ντεπρέ, σας ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικό και θα κάνετε και μια ερώτηση στην συγγήτρια. οπότε θέλετε να απαντήσετε. Να μιλήσω ισπανικά εγώ. Το μικρόφωνο της ε, ομιλήτρες δεν ήταν ανοιχτό, τώρα είναι, οπότε είναι εντάξει. Στην ε, έκθεση δυσκολευόμασταν πολύ στην πρώτη έκθεση για να κατανομάσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Φανταστείτε σε τι κατάσταση βρισκόμασταν τότε αν έπρεπε να μιλάμε για θύματα τρομοκρατίας ή όχι. Στην έκθεση που έγινε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, βάλαμε τελικά 31 τροπολογίες ε, με τις ανάγκες των θυμάτων. Και μιλήσαμε για την υπευθυνότητα, για την εναρμόνιση, όπως ε, είπαμε και εδώ. Στην αναθεώρηση αυτή, στην εφαρμογή αυτή, εννοείται ότι θα ζητήσουμε να υπάρχει εξασφάλιση ότι χωρίς διακρίσεις αντιμετωπίζονται οι ανάγκες όλων ε, των θυμάτων. Το ότι κάθε χώρα θα βάζει το ίδιο ποσό χρημάτων, αυτό είναι δύσκολο να το πετύχουμε. Αλλά ίσως να πούμε να υπάρχει ένα ελάχιστο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει η κάθε χώρα. Ένα ταμείο με κάποιο εγγυμένο ποσό για αυτές τις περιπτώσεις ίσως δεν θα ήταν κακή ιδέα. Θα το στηρίζαμε. Ευχαριστούμε για τη στήριξή σας. Περνάμε στο δεύτερο πάνελ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο δεύτερο πάνελ λοιπόν που έχει να κάνει με την προστασία και τη στήριξη των θυμάτων και με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω εδώ την δόκτωρα Μύρια Βασιλιάδου που είναι συντονίστρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα που έχουν να κάνουν με τη λαθροδιακίνηση και την εμπορία. Παρακαλώ, 10 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ που με καλέσατε και ευχαριστώ που ε, επανειλημμένα το Κοινοβούλιο ασχολείται και επιμένει ε, να ασχολείται με αυτό το ζήτημα γιατί είναι σημαντικό. Ε, να πω πρώτα ότι το, το πεδίο είναι πολύ ευρύτερο σε σχέση με την οδηγία για την καταπολέμηση εμπορία ανθρώπων, αλλά είναι αλληλένδετα τα ζητήματα στην εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει μια παρεμφερή προσέγγιση. Τώρα το καινούριο σε αυτή την οδηγία ήδη από το 2011 είναι ότι ζητάει ανεφόρον ε, προστασία ε, σε αρρωγή και προστασία για τα πρόσβαση πρόταση για τα, για τα θύματα. Ε, επειδή ασχολούμαστε και με τα θέματα της συμμόρφωσης, ε, της οδηγίας ε, για την εμπορία, θα ήθελα να αναφερθώ και στην έκθεση πρόοδου του 2016 από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, παρότι μπορεί να επαναλαμβάνω τα ίδια, νομίζω που έχετε ακούσει, νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι πρόκειται για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, της χάρτας των δικαιωμάτων. Έτσι, πρόκειται για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και επίσης είναι εξαιρετικά επικερδής ε, δραστηριότητα οργανωμένης εγκληματικότητας. Και όταν μιλάμε για αυτό, τι μιλάμε για αγοραπολισίες ανθρώπων για την εκμετάλλευσή τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουμε κατά συζητάμε αυτό το θέμα. Ε, είναι ποια είναι αυτά τα θύματα. Στην περίπτωση τη εμπορία, ε, πάνω από τα δύο τρίτα των θυμάτων είναι γυναίκες και κορίτσια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε αυτό, γιατί πέφτουν θύματα σεξουαλική εκμετάλλευση. 21% ε, για την εκμετάλλευση στο τομέα τη εργασία και υπάρχουν και διάφορε άλλε μορφέ εκμετάλλευσης. Θέλω να τονίσω επίση ότι το 2016 ο, ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστευσής εντόπισε 11.000 ε, κορίτσια και ε, γυναίκε που ήρθαν μέσω τη Λιβύης και τη Ιταλία από την Ιγυρία και το 80% έπεσαν θύματα εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση. Αυτά μόνο μέσα σε ένα χρόνο. 600% αύξηση από το 2014 ε, μέχρι σήμερα. Να, όταν μιλάμε για τα θύματα, ε, να θυμόμαστε αυτά τα, ε, αυτούς τους αστρονομικούς αριθμούς ανθρώπων που υποφέρουν και μην ξεχνάμε ότι διαρκώς διωγγώνεται το φαινόμενο. Όπως είπαμε για τις εποχιακούς εργαζόμενους, γιατί το αναφέρατε και εσείς αξιότιμη βουλευτά, ε, όντως πρόκειται για υπηκός από την Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ολλανδία, Ολλανδία, την Ουγγαρία και την Πολωνία. Δεν είναι μεταναστευτικό φαινόμενο, ε, αμυγός μεταναστευτικό φαινόμενο, αλλά δυστυχώς ε, είναι πολύ ευρύτερο. Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα θύματα είναι στο τέλος, δηλαδή είναι αργά για να γίνει κάτι. Ε, δεν υπάρχει θύμα εμπορίας ε, που, ε, να, όπου να μην εμπλέκονται χρήματα, αγοραπολισίες και χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούνται τα θύματα και ισχύουν οι κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης. Και συμφωνώ με τους βουλευτές ότι η πρόκληση είναι η εφαρμογή και όχι το ίδιο το νομοθέτημα. Το νομοθέτημα είναι ευρύτατο καινοτόμο, μελλοντοστραφές ε, και όντως ε, χρονολογείται εδώ και 8 χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν μελλοντοστραφές και ρηξικέλευτο ήδη τότε. Ε, έχουμε την έκθεση όπου εκτιμούμε την μεταγραφή της οδηγίας αλλά όχι την εφαρμογή της. Οπότε η εφαρμογή είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά για τα θύματα και με αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι προκύπτει από την έκθεση ε, πως έκαναν τα κράτη-μέλη σημαντικές προσπάθειες, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και θα ήθελα να τονίσω κάτι σε σχέση με την ε, άνευ όρων, αρρωγή και υποστήριξη για τα θύματα. Όχι να είναι συνάρτηση της βούλησης του θύματος να μετάσχει ε, στην έρευνα, τη διερεύνηση του, την διαλεύκανση του εγκλήματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι έχουμε μια πλατφόρμα ευρωπαϊκή με πάνω από 100 μη κάπα που εμπλέκονται για αυτό το ζήτημα και είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι τα θύματα ε, τα ε, συμφέροντα των θυμάτων είναι στον πυρήνα αυτού του πλατφόρμα και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους. Ε, σε αυτή την πρώτη έκθεση προοδεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πήρε τις πληροφορίες και από τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και τι λένε και αυτό το παραθέτουμε μέσα στην έκθεση είναι πως οι προκλήσεις που εντοπίζονται, ε, δηλαδή ε, εντοπίζονται τα παιδιά, τα ως ε, θύματα εμπορίας ανθρώπων. Ε, δεν ε, συντρέχουν όμως οι προποθέσει για να βρούμε κατάλληλα προσαρμοσμένες λύσεις ότι η πλειοψηφία των θυμάτων δεν ταυτοποιούνται και άρα δεν έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά τους. Αυτά είναι θεμελιώδη σημασία. Ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε συστήματα αποζημίωσης, δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις υποδοχής και αρρωγής που να προσαρμοσμένες σε ε, απαιτήσει ε, των εμφυλού χαρακτήρα. Ε, και ε, φυσικά ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να αναλάβουν δράση, αλλά αυτή είναι η κατάσταση και επίσης με εμπορία ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το αποτέλεσμα, συγγνώμη, ήταν το αντικείμενο μιας σύντομης ανασκόπησης του 2016 και 2017. Έχουμε μελέτη για ομάδες υψηλού κινδύνου για τα παιδιά, παραδείγματο χάρη δημοσιεύσαμε μαζί με το ΦΡΑ, τον Οργανισμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τα θέματα ό,τι σχετίζεται με τα θέματα κυδαιμονίας ε, για τα παιδιά. Επίσης, ε, αναγνώριση ταυτοποίηση των θυμάτων τη εμπορία ανθρώπων. Έχουμε πλέον ένα κατάλογο των θυμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για τα έμφυλα ζητήματα μελέτη που δημοσιεύσαμε. Το, τονίζουμε διαρκώς την σημασία να υπάρχουν υπερεθνικοί μηχανισμοί παραπομπή των ζητημάτων, ώστε να προσφέρεται η στήριξη στα θύματα. Είναι μέγιστη η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Επίσης, ε, χρηματοδότηση ε, συστημάτων συνεργασίας ε, για τέτοια διεθνικά συστήματα παραπομπής των φακέλων. Επίσης, δημοσίευση με τις νέε προτεραιότητε. Έχουμε κάνει πάρα πολλά και μία από τις τρεις βασικέ προτεραιότητε μας είναι ακριβώς να παράσχουμε καλύτερη πρόσβαση και να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των θυμάτων της εμπορίας. Φυσικά, Σύντομα θα παρουσιάσουμε στο Κοινοβούλιο την ε, δουλειά που έχουμε κάνει, αλλά το σημαντικό στην ανακοίνωση αυτή είναι να κάνουμε τα βήματα που χρειάζονται, ούτως ώστε να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να αναγνωριστούν ως κατοχή δικαιωμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ούτω ώστε να ε, ξεκαθαρίσουμε ότι έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δικαιώματα, να μεριμνήσουμε, ούτω ώστε να προστατευτούν και να διαφυλαχθούν αυτά τα δικαιώματα. Θα ήθελα να κλείσω τώρα λέγοντα και κάποια λόγια για το, την νομοθεσία. Είναι καλή ε, η νομοθεσία και ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων για τη φιλόδοξη αυτή νομοθεσία και έχουμε δεσμεύσει από πλευρά των κρατών μέλων. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλα αυτά. Προς το παρόν δεν υπάρχει όμως ορθή εφαρμογή και πρέπει να το τονίσουμε και το επαναλαμβάνουν και οι ευρωβουλευτές. Είναι αργά για τα θύματα. Πρέπει πραγματικά να... Όταν φτάνουμε στο επίπεδο του θύματος είναι αργά. Πρέπει να λειτουργήσουμε για την ε, πρόληψη. Είναι αστρονομικά τα ποσά, τα κέρδη της εμπορίας ε, ανθρώπων ε, και έχουμε μια περιγραφή των εθνικών νομοθετημάτων για την ποινικοποίηση των υπηρεσιών των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και των μέτρων που έχουν θεσπιστεί. Και τι βλέπουμε από αυτή τη μελέτη είναι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ε, αν χαρτογραφήσουμε αυτές τις νομοθεσίες ε, και καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει θύμα αν δεν υπάρχει ε, χρήστης, εκμεταλλευτής κέρδος. Και σε διάφορα κράτη-μέλη δεν ποινικοποιείται η αγορά των υπηρεσιών ακόμη και αν ξέρει κάποιος ότι πρόκειται για θέμα εμπορίας ε, ε, ανθρώπων. Δηλαδή, όταν υπάρχει αυτή η γνώση, παρόλα αυτά δεν με κοινοποιείται η αγορά των υπηρεσιών. Δεν υπάρχει νομοθεσία γι' αυτό και το κ. Σαβραμόπουλος ε, ε, είπε ότι δεν θα πρέπει να υποθάλπουμε αυτή την, αυτό το, το, πνεύμα ατιμορρησίας. Αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε και αυτό τονίζουμε στην ανακοίνωση του, 2000, του Δεκεμβρίου και νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανείς ότι αυτή, αυτή αυτό το πνεύμα τιμωρησία ε, πρέπει να ε, εκλείψει, διότι έχουμε χρηματοδότηση, έχουμε πολιτικές, έχουμε νομοθεσία και για να τους προστατεύσουμε, να τους ε, βοηθήσουμε, να φροντίσουμε να επανενταχθούν σε όλα αυτά τα στάδια της μακάβριας αυτής, απάνθρωπης αλυσίδα, εμπορία ανθρώπων. Το βασικό τρόπο που έχουμε να κάνουμε είναι να εμποδίσουμε αυτές τις αξιόπινες πράξεις και σας ευχαριστώ ειλικρινά που μας επικουρείται σε, αυτό το μας το εγχείρημα. Σας ευχαριστούμε κυρία Βασιλιάδου. Τώρα ο κύριο Χαβιέζας Μπάντα, ερευνητής ε, που εμπλέκεται σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα για τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών. Παρακαλώ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα επικεντρωθώ σε δύο θέματα. Πρώτον, θα σας μιλήσω για τον τρόπο με τον οποίο μεταχειριστήκαμε τα θύματα τρομοκρατίας στη χώρα των Βάσκων και μετά θα σας μιλήσω για τη βασική ανάγκη δικαιοσύνης. Αυτό ζητούν τα θύματα ακριβώς για να θυμόμαστε τα θύματα αυτά, ζητούν δικαιοσύνη. Στην περίπτωση λοιπόν της χώρας των Βάσκων και της Ισπανίας γενικότερα, όπως γνωρίζετε, είχαμε τρομοκρατία για πολλά χρόνια, πάνω από 50 χρόνια η οποία κατέληξε σε πάνω από 800 θύματα και βέβαια σε πολύ μεγάλη οικονομική ζημιά. Πώς βοηθήθηκαν τα θύματα αυτά τρομοκρατία στη ΣΕΤΑ στη χώρα των Βάσκων. Όταν πλησιάζουμε τα θύματα τρομοκρατίας πρέπει να ξέρουμε ότι έχουν υποστεί την τρομοκρατική ενέργεια, άρα έχουν περάσει από μια τραυματική εμπειρία γιατί έχουν χάσει τους δικούς τους ή έχουν τραυματιστεί. Οπότε πέρασαν από αυτό το κίνδυνο, από αυτή την τραυματική εμπειρία από την οποία κινδύνευσε η ζωή τους, η φυσική τους ακεραιότητα. Είναι κάτι έκτακτο στη ζωή τους. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις ουσιαστικά πλήττει την εμπιστοσύνη του ανθρώπου στην καθημερινότητό του. Πάβει να νιώθει ασφαλής και αυτό είναι κάτι από... πάρα πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην καθημερινότητα. Και είναι κάτι που δεν περιορίζεται στις ηλικέ απώλειες, είναι έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στους συνανθρώπους και στον ίδιο μας τον εαυτό. Υπάρχουν ε, μελέτες για τις ψυχολογικές επιπτώσεις της τρομοκρατίας στα θύματα. Όσοι υποφέρουν λοιπόν από αυτού του είδους ε, τρομοκρατικές επιθέσεις χρειάζονται μια ειδική στήριξη και πολύ συγκεκριμένη, πολύ ειδική. Γιατί η ζωή τους θα βασιστεί στην κοινωνική στήριξη, την ε, στήριξη των συγγενών και στην αποκατάσταση της υγείας του της ψυχολογικής και της σωματικής. Είναι τραυματική εμπειρία όπως είπαμε. Είναι ένα τραύμα, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό και πρέπει να το ξεπεράσουν τα θύματα. Γι' αυτό και η κοινωνία έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει απέναντι στα θύματα. Χρειάζεται αλληλεγγύη, κοινωνική στήριξη. Είναι πολύ βασικό, βοηθάει πολύ τα θύματα. Θέλω επίση εδώ να αναφερθώ στην τρομοκρατία της ΕΤΑ. Ήταν κάτι πολύ βασικό στην ιστορία της Ισπανίας και επεκτάθηκε και στην Ευρώπη. Εμείς 50 χρόνια λοιπόν υποφέραμε ως ισπανική κοινωνία από την τρομοκρατία αυτή και ειδικότερα βέβαια η χώρα των Βάσκων. Η πραγματικότητα που ζήσαμε με την τρομοκρατία τη ΣΕΤΑ στη χώρα των Βάσκων ήταν μια πολύ ιδιαίτερη πραγματικότητα γιατί τα θύματα ω επιτοπλίστων στη χώρα των Βάσκων Τη μόνη στήριξη που είχαν ήταν το συγγενών τους και των φίλων τους. Για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι πολύ πρόσφατα, δεν είχαν τίποτα άλλο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούνε στήριξη εκτός από το στενό οικογενειακό κύκλο. Γι' αυτό τα θύματα της τρομοκρατίας στη χώρα των, Βίσκο, των Βάσκων ε, κατέστησαν διπλά και τριπλά θύματα. Χρειάζεται κοινωνική ε, υποστήριξη πολλές φορές δόθηκε το όνομα του θύματος που έχασε τη ζωή του στους δρόμους και το ότι η κοινωνία ε, της χώρας των Βάσκων έδειξε πως συμπάσχει με το θύμα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τα θύματα. ως θύματα της τρομοκρατίας με τη στήριξη της κοινωνίας κατάφεραν να ξεπεράσουν κάπως αυτό το καθεστώς του θύματος. Πολλοί είδαν να δολοφονούνται οι γονείς τους. Και το τραύμα αυτό του ακολουθεί σε ολόκληρη τη ζωή τους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η μελέτη για το πώς αντιμετώπισε η κοινωνία της χώρας των Βάσκων την τρομοκρατία εκεί. Με αδιαφορία από το κράτος καταρχήν. Και τι έγινε όμως με αυτούς οι οποίοι ήταν οι θήτες οι οποίοι κατέληξαν στη φυλακή. Εδώ θα σας έλεγα τρία πράγματα τα οποία θα έπρεπε να φροντίσουμε. Το ένα είναι ο σεβασμός. Τι σημαίνει σημαίνει να ξεχάσουμε την πολιτική ή τη θρησκευτική διάσταση. Πρέπει να δείξουμε ότι συμπάσχουμε, να χρησιμοποιήσουμε τη σωστή γλώσσα. Είναι πολύ σημαντική γλώσσα που χρησιμοποιούμε και που δεν το φροντίσε πάντα η αρμόδια υπηρεσία της χώρας των Βάσκων. Μερικές φορές, και πολλές μάλιστα, η γλώσσα που χρησιμοποιείται δεν είναι η γλώσσα της αλήθειας το πώς έγιναν ακριβώς τα πράγματα. Προσπαθούν να μετριάσουν κάπως. Χρησιμοποιείται μία γλώσσα η οποία δεν δέχεται το τι πραγματικά έγινε. Ε, προσπαθούν να είναι πολιτικά ορθά τα λόγια τα οποία εκφέρουν πολύ ε, Μιλούν για θανάτους αντί να μιλούν για δολοφονίες, για παράδειγμα. ή μιλούν για δολοφονίες, δεν μιλούν για εκτελέσεις. Πώς θα προσεγγίσει κανείς ένα θύμα τρομοκρατίας στη χώρα των Βάσκων είναι πιο δύσκολο από ότι είναι αλλού στην Ισπανία ή αλλού στην Ευρώπη. Γιατί υπάρχει πάντα αυτή η κοινωνική διάσταση στη χώρα των Βάσκων που μερικές φορές στηρίζουν την τρομοκρατία. Οπότε είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση των θυμάτων εκεί. Πρέπει κανείς με ειλικρίνεια και ευαισθησία να πλησιάσει το θύμα, να καταλάβει τι έχει υποφέρει, ότι έχει πίσω το ένα μεγάλο τραύμα. Και όταν η κοινωνική στήριξη μάλιστα είναι μηδενική, καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για το θύμα και έτσι είναι στη χώρα των ε, Βάσκων. Τέλος θέλω να μιλήσω για την ανάγκη δικαιοσύνης όσον αφορά τα θύματα τρομοκρατίας αλλά και άλλων εγκληματικών εργειών Συγκεκριμένα στη χώρα των Βάσκων τα θύματα ξέρουν ότι δεν υπάρχει νόμος για να τους βοηθήσει. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη αποκατάστασης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει και τίποτα. Σε διεθνές επίπεδο πολλοί ασχολούνται με αυτά αλλά δυστυχώς ακόμα επειδή υπάρχει η ιδέα της προστασίας των ε, καταδικασμένων, των δικαιωμάτων τους κτλ. Τελικά μερικές φορές καταλήγουν σε ατιμορρησία. Πρέπει να ξέρουμε ότι η τρομοκρατία και κυρίως τη ΣΕΤΑ ήταν κάτι το οποίο δεν πέρασε ουσιαστικά από καμία τιμωρία, δεν προσφέρθηκε καμία αποκατάσταση στα θύματα. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Εμείς πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ίδια για όλα τα θύματα. Τα θύματα έχουν το ηθικό δικαίωμα να πετήσουν δικαιοσύνη και αυτό είναι πολύ βασικό. Πρόσφατα αναγνωρίστηκε και από την Μάρτα Ρικένα που είναι η Διευθύντρια της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την Τρομοκρατία. Και στον ΟΗΕ είχε ακουστεί ότι εδώ πέρα πρόκειται για μια ολόκληρη κοινωνία που πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην οδηγία αυτή του 2012 αναγνωρίζει την ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα θύματα τρομοκρατίας απέναντι στη δικαιοσύνη. Χρειάζεται δικαιοσύνη για τα θύματα και μιλάω εδώ για τις 370 δολοφονίες της ΕΤΑ που δεν έχουν επιληθεί ακόμα. Ούτε 40% των ε, δολοφονιών της ΕΤΑ. Οι μισές περιπτώσεις δηλαδή δολοφονιών της ΕΤΑ δεν έχουν ε, διευκρινιστεί. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να συλλεχθούν στοιχεία και να υπάρξει δικαιοσύνη. Χρειάζονται αποτελεσματικά εργαλεία. Δεν είναι δυνατόν να έχουν μείνει τόσε περιπτώσει αδιευκρίνηστε. Χρειάζεται συνεργασία με τι αστυνομικέ και άλλε αρχέ, με δημοσιογράφου, Θέλουμε να υπενθυμίσουμε και τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης του Δεκεμβρίου του 1996 που μίλησε για την καταπολέμηση των εγκλημάτων των, ε, του οργανωμένου εγκλήματος και έκανε συστάσεις για την αποτελεσματική ε, διελεύκανση των εγκλημάτων αυτών με αναλογικότητα. Το σύστημα ελευθεριών μας θέλουμε να τιμωρεί τους τρομοκράτες και τους συνενόχους τους και όχι το αντίθετο. Τέλος, πρέπει να επιμείνουμε ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οριστική ειρήνη στην Ισπανία και στη χώρα των Βάσκων κυρίως, αν οι τρομοκράτες δεν εκτίσουν πλήρως τις ποινές τους και αν δεν διαλευκανθούν και τα εγκλήματα αυτά τα οποία παραμένουν χωρίς να έχουν επιληθεί. Γι' αυτό πρέπει να ακούσουμε τα θύματα και τους εκπροσώπους τους. Τα θύματα της τρομοκρατίας, της ολοκληρωτικής τρομοκρατίας, πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να προστατευτούν γιατί η τρομοκρατία δεν σταματάει. Ευχαριστούμε πολύ. Ο δόκτωρ Κεβάτ είναι τώρα, καθηγητής συγκριτικού δικαίου και νομικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο του Τούρκου. Παρακαλώ, μπορώ να έχω τις διαφάνειες. Thank you. And thank you for the for... Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει πάρει τόσο ζεστά το θέμα των θυμάτων ε, της τρομοκρατίας. Προσπαθώ να καλύψω εδώ πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, προσπαθώντας να περιγράψουμε τα νομικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για τα δικαιώματα των θυμάτων και μετά θα συζητήσουμε ευρύτερα πώς εφαρμόζονται αυτά. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε περάσει από μια τεράστια εξέλιξη όσον αφορά το ποινικό δίκαιο. Πριν από μερικές δεκαετίες η ιδέα ήταν ότι το κράτος έπρεπε να τιμωρεί τους δράστες και να προστατεύει τα θύματα. Τώρα έχουμε διαφορετική στάση απέναντι στις ποινικέ διαδικασίες και το ποινικό δίκαιο. Και όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τώρα Προσπαθούμε βέβαια να έχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των θυμάτων και τα δικαιώματα των θητών. Παρ' όλα αυτά υπάρχει η συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 82, έχουμε την νομική βάση για τα θύματα και τους θύτες. Ακόμα δηλαδή τα θύματα δεν βρίσκονται στο κέντρο της διαδικασίας. Προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία. Πρέπει να δούμε ποια είναι η δικαία όμως, η δίκαια όμως ισορροπία. Τι σημαίνει μια δίκαια δίκη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό όταν μιλάμε για ευάλωτα θύματα. Τότε η ισορροπία κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι διαφορετική. Τώρα λοιπόν μιλάμε για την οδηγία για τα θύματα. Πρόκειται για ένα νομικό μέσο προκειμένου να βελτιώσουμε τα δικαιώματα των κοινών θυμάτων, ας πούμε, αλλά γίνεται μνήα και στα ευάλωτα θύματα στην οδηγία αυτή. Από την άλλη, έχουμε μία σειρά νομικών εγγράφων, τα οποία επικεντρώνονται σε διάφορες ομάδες θυμάτων. Και όλα αυτά τα θέματα έχουν τις ρίζες τους σε πολιτικές, για ευάλωτες ομάδες και για τέτοιες καταστάσεις όπου κάποιες ομάδες ανθρώπων πραγματικά έχουν γίνει ευάλωτες λόγω του καθεστώτος τους και των ε, σχέσεών τους με τους θύτες και τους έχουν αρνηθεί τα δικαιώματά τους. Να σας υπενθυμίσω ότι όταν μιλάμε για βάλωτες ομάδες θυμάτων, οι θύτες απείλαυσαν νομική de facto ατιμορρησία έναντι του ποινικού δικαίου. Αυτή είναι η παράδοση ε, που αντιμετωπίζουμε. Άρα υπήρξε πολύ αργή ε, νομική αναγνώριση κατά αυτών των πράξεων, κατά των ευαλώτων ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν καταγγελθεί επαρκώς τα εγκλήματα, δεν έχουν γίνει οι διώξεις όπως έπρεπε και δεν έχουν επιβληθεί κατάλληλες κυρώσεις και αυτό συνεχίζεται. Απ' την άλλη βέβαια τα θύματα φοβούνται τον θήτη, πολύ συχνά έχουν περιορισμένη δυνατότητα να δράσουν και αυτό παρεμποδίζει την καταγγελία των εγκλημάτων. Μπορώ να πω ότι εργάστηκα πολύ πάνω σε αυτά τα ζητήματα για την παροχή βοηθείας σε θύματα ε, σεξουαλικής βίας και άλλα παρέμφερη. Και το θέμα αφορά κυρίως το φόβο, πάρα πολύ το φόβο. Τι γίνεται άμα καταγγείλεις ένα έγκλημα. Ευάλωτα θύματα πρέπει να αναγνωριστούν. Το χρειάζονται αυτό. Και χρειάζονται και υπηρεσίες στήριξης. Ε, επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Ε, έχουμε δύο ομάδες οδηγιών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Από τη μία πλευρά έχουμε την οδηγία για τα θύματα, εκεί καθορίζονται τα ευάλωτα άτομα ή που πρέπει να θεωρούνται ευάλωτα θύματα και μετά έχουμε ομάδα οδηγιών με ε, κάλυψη συγκεκριμένων καταστάσεων και είδη αδικημάτων και εγκλημάτων, όπου η οδηγία για την σεξουαλική ε, ε, παρενόχληση των παιδιών, θέματα, θύματα τρομοκρατίες κλπ. Και αυτά τα δύο είδη εργαλείων είναι διαφορετικά. Την επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Η εφαρμογή λοιπόν, αυτή η αξιολόγηση μάλλον, για την υλοποίηση των μέτρων ε, θέτει το θέμα κατά πόσο θα πρέπει να, ληφθεί υπόψη αυτή η πτυχή σε όλα τα νομικά εργαλεία που διαθέτουμε. Βασικά οι οδηγίες για την ε, βιοπραγία κατά των παιδιών και την τρομοκρατία κλπ. είναι εργαλεία του ποινικού δικαίου. Το ίδιο ισχύει και για τη βία κατά των γυναικών σε πολλές περιπτώσεις, επί παραδείγματι, υπάρχει σαφής ανάγκη σε αυτή την περίπτωση να γίνει κάτι για αυτά τα εγκλήματα. Τι σημαίνει, τι συμβαίνει τώρα βάσει των μέσων αυτών, των εργαλείων αυτών. Χρειάζεται το κίνητρο για την καταστολή του εγκλήματος υπερτερεί της ανάγκης προστασίας των θυμάτων. Αυτό πρέπει κάπως να λαμβάνεται υπόψη όταν αυτές οι πτυχές ενσωματώνονται σε άλλες πολιτικές ε, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να πω κάποια πράγματα για διάφορα θέματα που άπτονται της αναγνωρίσεως των ευαλώτων θυμάτων. Ίσως μπορούμε να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού όσον αφορά τους διάφορους φορείς που εμπλέκονται. Ε, αυτό ε, εξαρτάται από το ότι οι ΜΚΟ πολύ συχνά ε, δραστηριοποιούνται όταν τα κράτη αδρανούν. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα μεγάλο όσον αφορά την πρόσβαση στις υπηρεσίες. Και αυτό είναι πολύ κακό σε περίπτωση των ευαλώτων θυμάτων. Ε, που πρέπει να υπάρχει ένα σαφέστατο πρότυπο και είναι σαφές από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή ότι ο συντονισμός των προσπαθειών είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να επιληθεί από το κράτος. Είναι σαφέστατο αυτό. Δεν θα πρέπει να το αφήνουμε ε, να κινείται από μόνο του, να ανατίσσεται από μόνο του. Επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, η μία επαρκή καταγγελία εγκλημάτων. Η ανελειπή καταγγελία. Συγγνώμη, η ελλειπής καταγγελία εγκλημάτων. Αυτό είναι κάτι που διαπιστώνεται επανειλημμένα. Ότι αυτή η ελλειπής καταγγελία είναι μεγάλο πρόβλημα και αφορά τα ευάλωτα θύματα. Και αυτό οφείλεται εν μέρη στο γεγονός ότι οι χώρες κατά κάποιο τρόπο έχουν αναθέσει σε άλλους την προστασία των ευαλώτων θυμάτων, δηλαδή σε ο Καλό αυτό σε πολλές περιστάσεις. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με την πρώτη επαφή. Εκεί γίνεται με τα, αυτούς που είναι επανειλημμένα θύματα και συναντούν άλλους ε, το, τις αγγελικές αρχές, την αστυνομία κλπ τι γίνεται σε αυτές τις περιστάσεις. Χρειάζεται ε, ε, δημιουργία ενός σημείου εισόδου για αυτούς τους ανθρώπους, για να σε επαφή με τις αρχές. Επόμενη διαφάνεια. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο είναι σημαντικό να πούμε ότι θα πρέπει κανείς να δρά εξοφίσιο, δηλαδή αυτεπάγγελτα να γίνονται οι παραπομπές και οι καταγγελίες κλπ. Να γίνει βασικός ε, κανόνας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα ευάλωτα θέματα. Η αυτεπάγγελτη κίνηση των διαδικασιών. Ευχαριστώ πολύ, Δόκτωρ Νουσιάνεν. Και τώρα, επόμενος ομιλητής, η κυρία Ελίζα Μπεθράουλετς, επικεφαλής της ΥΜΕΑ της Υπηρεσίας Διαμορφώσεως Πολιτικής και της Task Force για τις πρωτοβουλίε για τα δύο φύλλα και το εκπρόσωπο του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ήθελα να μας μιλήσει η κυρία Κάουλετς ε, στι ε, στις προσωπικές εμπειρίες αθήμα της τρομοκρατίας. Σας καλωσορίζουμε. Σας εκφράζουμε την υποστήριξή μας και έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωκοινοβούλιο και αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις ε, που έχουν στο θεματολόγιο αυτό το σημαντικό θέμα. Δύο χρόνια μετά την τρομοκρατική επίθεση του Ζάβεντεμ το αυτό, Διότι ήμουν στο Ζάβεντεμ στις 22 Μαρτίου του 2016 και δύο χρόνια αργότερα σχεδόν αισθανόμαστε ότι έχει ξεχαστεί σχεδόν αυτή η υπόθεση. Να σας δώσω ένα-δύο παραδείγματα για το αισθάνομαι αυτό. Είμαι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μένω στις Βρυξέλλες. Για πάνω πέντε χρόνια μένω στις Βρυξέλλες και είμαι από την Ουγγαρία. Η κόρη μου είναι νέα ετών και πειράστηκε άμεσα, επλήγει άμεσα από αυτό που συνέβη. Άκουσα σήμερα ότι θεωρούμε θύματα του συγγενείς ε, που ε, εξετάζουμε τι γίνεται με τους συγγενείς των θυμάτων που πέθανα. Εγώ δεν πέθανα, αλλά η κόρη μου είναι ακόμα νέα και είναι πολύ δύσκολο ακόμα για εκείνη να ξεπεράσει την τρομοκρατική επίθεση. Είμαι πρώην διπλωμάτης, είμαι οικονομολόγος και εργάζομαι για την EUYS, e δραστηριοποιούμε και στην EMCHAM, γιατί είναι σημαντικό, διότι Αντί να παρετηθώ, αποφάσισα να επιστρέψω στην πραγματικότητα και την κανονικότητα το ταχύτερο δυνατόν. Αυτό επέλεξα. Και όσον αφορά τη στήριξη που έλαβα, χαίρομαι που άκουσα για την οδηγία και όλα αυτά που συμβαίνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αλλά αισθάνομαι ότι είναι πολύ σημαντικό να πω ότι όλη η υποστήριξη που έλαβα ήταν από την οικογένειά μου, από τους φίλους μου και από τους εργοδότες μου, την EY. Είμαι προγνώμων διότι ε, από άλλη πλευρά δεν είχα υποστήριξη. Πήγα στο νοσοκομείο για πάνω από τρεις εβδομάδες. Δεν ξέρω αν μπορεί να αποχωρήσετε με τις διαφάνειες. Δεν είναι επαγγελματικέ ε, φωτογραφίες και εικόνες. Απλώς κάποιες εικόνες δείχνω για να σας δείξω πώς μπορεί να αλλάξει ε, μια ανοιχτή ζωή κάποιου Η προηγούμενη εικόνα ήταν όταν ήμουν ακόμα στο νοσοκομείο και όταν ήθελα να με επισκεφτούν στο νοσοκομείο είχα υποστήριξη για τρεις εβδομάδες και ευχαριστώ τους γιατρούς, της νοσοκόμες, τους νοσοκόμους και όλους αυτούς που ήταν εκεί. Μετά από δύο εβδομάδες έφυγα από το νοσοκομείο, Ήμουν αμόνιμο μετά με το πρόβλημά μου και στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ότι είναι σημαντικό το θέμα. Όπως βλέπετε Τότε ζούσα σε ένα διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο, που είναι ουσιαστικά τρίτος όροφος, χωρίς ασανσέρ. Για τρεις μήνες δεν μπορούσα να φύγω από το διαμέρισμα χωρίς εξωτερική υποστήριξη. Και εξωτερική υποστήριξη ήταν ε, το νοσοκομιακό και οι φίλοι μου που ερχόταν από παντού να με επισκεφθούν και να με βοηθήσουν να με μεταφέρουν κάτω. με βοηθούσαν, μου κρατούσαν παρέα και μπορούσαν να με βοηθήσουν να ξεφύγω και από τον τρόμο που ήταν συνέχεια στο μυαλό μου. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ότι πρέπει να δείξουμε ότι στην περίπτωσή μου και υπάρχουν και άλλα θύματα πιστεύω γι' αυτό που αναφέρω δεν είναι θέμα αν ήμασταν θύματα ή όχι αλλά υπάρχουν στοιχεία και αστυνομία και όλοι γνωρίζουν τούτου λεχθέντος δεν έτυχα άλλη υποστηρίξους. Κανείς δεν προσήγησε να με ρωτήσει αν χρειάζομαι κάτι. Πήρα ένα email από επίτροπο για την υποστήριξη των θυμάτων και χάρηκα που έλαβα και ένα τηλεφώνημα. Στην πράξη όμως έλαβα ένα email με διάφορες σελίδες που έπρεπε να συμπληρώσω για να λάβω άμεση οικονομική υποστήριξη Προφανώς δεν ήμουνα σε θέση να συμπληρώσω όλα αυτά τα έγγραφα και τότε δεν έλαβα καμία οικονομική υποστήριξη Τότε των λεχθέτων στο αεροδρόμιο έχασα τα πάντα. Έχασα τις κάρτες μου, τις, τις πιστοτικές μου, άφησα τα πάντα εκεί. Και αυτό είναι το μόνο στοιχείο που βγήκε από τη βαλίτσα μου που καταστράφηκε. Και την στράφη χάρη σε μια φίλη που είναι στην αίθουσα. Μετά από εβδομάδες. Τα πάντα καταστράφηκαν. Οι κάρτες μου χάθηκαν. Ήμουν σε ξένη χώρα. Σαν μια μητέρα με την κόρη της. Χωρίς λεφτά στη τσέπη μου. Τίποτα. Χωρίς την υποστήριξη οικογένειας και συναδέλφων και φίλων δεν θα μπορούσα να επιβιώσω και να είμαι εδώ σήμερα. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό που θέλω να πω. Πολλοί από εσά και το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζουν διάφορα στοιχεία όπως και την οικονομική υποστήριξη. Μετά από δύο χρόνια σχεδόν δεν έχω λάβει την παραμικρή οικονομική υποστήριξη. Αυτό που πέρασα είναι ότι πέρασα πολλού πολλούς γιατρούς ασφαλιστικών εταιριών, πάνω από 10 γιατρούς πέρασα ασφαλιστικών εταιριών, κάθε φορά πέρναγα από τέσσερις γιατρούς εξηγώντα τι πέρασα και πέρναγα και ξανά και ξανά τον ίδιο τρόμο και τη φρίκη με το μυαλό μου και αυτό δεν με οδήγησε σε μια ανάκαμψη. Με επέστρεφα συνέχεια σε αυτό που συνέβη. Αυτό δεν με βοηθάει να το ξεπεράσω. Πάνω από δέκα γιατρούς, 10 επισκέψεις γιατρών των ασφαλιστικών εταιριών πέρασα. Κάποιες από τις εξετάσεις ήταν αρκετά δυνηρές. Μετά την πρώτη ε, ε, πέρασα από μια κρίση πανικού, διότι δεν σταματούσε ο γιατρός τις ερωτήσεις και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς υποβάλλονται οι ερωτήσεις δεν κατάλαβα γιατί μου έβαλα τους ερωτήσεις όλοι, ήξεραν ότι ήμουν εκεί, τραυματίστηκα και έμεινα στα χέρια των ασφαλιστικών εταιριών, των γιατρών των ασφαλιστικών εταιριών και ακόμα δεν πήρα δεκάρα. Οι ιατρικές δαπάνες καλύφθηκαν, αλλά είναι προφανές στη σπάση ότι ε, ήμουν επαγγελματής, ταξίδευα σε άλλη χώρα να συζητήσω σημαντικά θέματα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Διότι δεν έχω περισσότερο χρόνο και δεν θέλω να σας δώσω κάθε προσωπική πληροφορία. Όλοι όμως μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχουν πολλών άλλων ειδών απώλειες. Επαγγελματικά αυτή η απώλεια ήρθε την χείριστη στιγμή. Διότι έβγαινε στη σύνταξη το αφεντικό μου και ήλπιζα να πάρω κάποια προαγωγή. Δεν πήρα προαγωγή τότε και ακόμα ελπίζω ότι κάποια μέρα θα επιστρέψω στο σωστό μονοπάτι και θα πάρω την προαγωγή που ήλπιζα τότε να την πάρω σύντομα τώρα. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Παρακαλώ, ε, πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε το τραύμα. Να η κόρη μου και η οικογένειά μου Έχω και διάφορες άλλες εικόνες να σας δείξω ότι ήμουν πράγματι σαν απειρικό καρουτσάκι και οι γιατροί των ασφαλιστικών εταιριών το ήξεραν. Και παρόλα αυτά, τότε και σήμερα ακόμα, έπρεπε να σε αντιμετωπίσω. Στο εγγύς μέλλον, έχω άλλους τρεις γιατρούς ασφαλιστικών που πρέπει να συναντήσω και ακόμα δεν έχω πάρει οικονομική αποζημίωση. Η προηγούμενη διαφάνεια είναι μια εικόνα με τον πρόεδρο της Ουγγαρίας που με κάλεσε πολύ καλή χειρονομία και όλη η υποστήριξη που έλαβα ήταν υποστήριξη που έλαβα από την Ουγγαρία που είναι η χώρα μου. Με κάλεσε ο πρεσβευτής, με επισκέφτη μου προσέφερε να με μεταφέρει, να με επιστρέψει στην Ουγγαρία. Αυτό δεν ήταν όμως επιλογή για μένα. Γιατί? Διότι μένω στο Βέλγιο, είναι η κόρη μου εδώ. Ζω εδώ για πάνω πέντε χρόνια. Οπότε δεν μπορεί κανείς να επιστρέψει ξανά σε, σε άλλη χώρα. Στην πρώτη φωτογραφία, δεν σας λέω να πάτε πίσω, αλλά θα βλέπατε ότι ήμουνα στον πάνω όροφο, δεν μπορούσα να μετακινηθώ και έπρεπε λοιπόν να πάρω μια απόφαση, άμεση απόφαση, να μετακομίσω, να αγοράσω άλλο διαμέρισμα που να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση, να είναι κοντά στη δουλειά μου, κοντά στην κόρη μου, ένα διαμέρισμα πληρούσε όλα τα κριτήρια ε, και ήταν ε, πολύ περάνω των οικονομικών μου δυνατοτήτων, έπρεπε όμως να δεσμευτώ, να προσπαθήσω για να επιβιώσω και το δάνειο, πήρα δάνειο που έπρεπε να αποπληρώσω και έχω επηρεαστεί, έχω πληγεί οικονομικά. Και όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα είναι αποτέλεσμα της τρομοκρατικής αυτής πράξης. Κλείνοντας λοιπόν, στην παρέμβασή μου θέλω να πω τα εξή. Δεν θέλω να κάνω κάποιες συστάσεις. Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό. Τούτου λεχθέντος όμως, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποια πολύ εύκολα εργαλεία που θα μπορούσαν να με βοηθήσουν τότε. Πολλοί από εσά αναφερθήκατε στο ένα σημείο επαφής. Ένα ενίο σημείο επαφής θα ήταν απίστευτα σημαντικό. Ασφάλεια, αποζημίωση, νομική αρρωγή, όλες αυτές οι ευθύνες δεν θα πρέπει να βαρύνουν κάποιον που παλεύει να ξανασταθεί στα πόδια του και να επιστρέψει την πραγματικότητα πέρα από την φυσική ζημιά, τη σωματική ζημιά και η ψυχολογική ζημιά πρέπει να εξεταστεί και να θεωρηθεί εξίσου σημαντική. Αυτόματη αποζημίωση που θα βασίζεται σε στοιχεία, πραγματικά στοιχεία. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, αυταπόδεικτον αυτό, αυτονόητο. Μια προκαταβολή σε ρευστό δεν, απαιτεί, δεν πρέπει να απαιτεί συμπλήρωση κι άλλων εντύπων. Προφανώς κάποιο που υποφέρει σε νοσοκομείο δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και για μένα που είμαι ε, μια μέλος μονογονικής οικογένειας, ε, μια υποστήριξη όπως μια νοσηλεύτρια που θα με σκεφτόταν θα βοηθούσε. Η μητέρα μου ήταν μαζί μου και ήμουν πολύ τυχερή σε αυτό. Αλλά υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, άλλες γυναίκες για τις οποίες θα ήταν πολύ σημαντικό κάτι τέτοιο. Και πρέπει να το αναφέρει αυτό η Επιτροπή. Ευχαριστώ ξανά που κρατάτε ακόμα αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξή σας. Ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μαζί μας ε, ε, την προσωπική σας ιστορία και εκφράζουμε την ε, λύπη και κατανόησή μας για αυτή, αυτό που περάσατε. Θα περάσουμε τώρα στην ανταλλαγή απόψεων για να έχουμε και τις ερωτήσεις από τα μέλη. Η Άννα Χίτ. Δύο λεπτά. Γιατί στις 12.30 ακριβώς θα διακόψουμε διότι συνεδριάζουν οι συντονιστές. ε, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Σας ευχαριστώ για όλες ε, τις ε, πληροφορίες που μας δώσατε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία, λυπηρή και ιδιαίτερα σημαντικό που σας ακούσαμε. Ε, μία ερώτηση έχω μόνο προς την δόκτωρα Βασιλιάδου. που ε, μας μίλησε πολύ για την ε, εμπορία ανθρώπων. Είπε η Μίριμ ότι ε, τα κράτη-μέλη έχουν νομοθεσία από το 2011, την έχουν μεταφέρει όμως νομοθεσία με πολύ διαφορετικό τρόπο και είναι πολύ δύσκολο γιατί χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, έχεις κάποιες σκέψεις, κάποιες προτάσεις, ιδέες, πώς μπορούμε να μεριμνήσουμε ούτω ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συγκρισιμότητα και ομοιότητα κατά τη μεταφορά της νομοθεσίας. Επίσης, ε, ακούστηκαν για κάποιες ιδέες ότι ίσως χρειαζόταν αναθεώρηση ε, της νομοθεσίας και ίσως πρέπει να ε, κινηθούμε λίγο νωρίτερα από ό,τι ε, ήθιστε, ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά και η εφαρμογή τη νομοθεσία γίνεται με πάρα πολύ διαφορετικό τρόπο, γιατί μας μιλήσει για την εφαρμογή. Ευχαριστούμε ο κύριος Ντεπρέ και η κυρία Γκόμες. Κύριο Ντεπρέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με άγγιξε πολύ η μαρτυρία του θύματος που μόλις ακούσαμε. και ε, αυτή την ε, χρονική στιγμή φάνηκαν τα κενά που υπάρχουν στη χώρα μου. Ε, δεν ήμασταν έτοιμοι. Ήταν ευνίδιο, δεν ήμασταν έτοιμοι, το παραδεχόμαστε και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και μεταξύ άλλων αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ένα ενιαίο σημείο επαφής. Αυτό ήδη λειτουργεί τώρα. Για τα θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα, παρακολούθηση, όλες, όλα τα έξοδα, τα έξοδα που δεν καλύπτονται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Ζητώ λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχει βοήθεια προς τα κράτη-μέλη ώστε να εναρμονιστούν οι διατάξεις για τα οικονομικά μέσα που μπορούν να κινητοποιηθούν για να ε, βοηθήσουμε τα, θύματα για να έχουν την κατάλληλη περίθαλψη, αλλά όχι μόνο, αλλά και στις διάφορες τομείς της ζωής τους να έχουν μια υποστήριξη ε, για την ε, μετατραυματική υποστήριξη, παραδείγματος χάρη την ψυχολογική υποστήριξη αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστούμε, Άννα Ε, θα ήθελα ευχαριστήσω ε, το θύμα της ε, τρομοκρατικής επίθεσης που μοιράστηκε την ιστορία της μαζί μας. Σχεδόν το μισό του χρόνου μου το περνάω στις Βρυξέλλες και νιώθω και ότι με αγγίζει προσωπικά αυτή η δοκιμασία που πέρασε η φίλη μας από την Ουγγαρία. Εγώ είμαι Πορτογαλίδα. Εμεί έχουμε τρομακτικές πυρκαγιές. Ε, είχαμε το, το, το καλοκαίρι. Πάνω από 100 άνθρωποι πέθαναν. Ε, πάνω από 200 τραυματίες είχαμε. Και το, αυτό που μου λένε τα θύματα είναι ότι πόσο σημαντικό ήταν για τους ε, επιζώντες να έχουν ε, ψυχολογική ε, υποστήριξη και κάτι που προσφέρουν οι πορτογαλικές αρχές. Και μου έκανε εντύπωση που ε, αναφέρατε ότι μια νοσοκόμα αν ερχόταν θα ήταν εξίσου σημαντικό με την υποστήριξη οικονομική για σας, για το παιδί σας. δεν, δεν, ότι, ε, δεν ότι χρειάζεται και η ψυχολογική υποστήριξη τα θύματα στην Πορτογαλία, γιατί τα Χριστούγεννα, παραδείγματος χάρη, έλεγαν πόσο απαραίτητο ήταν αυτό για να ε, δεχτούν τις απώλειές τους και τα θύματα και ε, έχασαν μέλη της οικογένειάς τους και χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη για να προσφερθεί αυτή όμως, να παρασχεθεί αυτή χρειάζεται προετοιμασία. Δεν χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε μια ειδική σύσταση για ψυχολογική υποστήριξη. Δεν χρειάζεστε ε, κάτι τέτοιο, κυρίως όταν μιλάμε για θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων. Χιμένες Μπεσερίλ. Ευχαριστώ. Το άλλο μικρόφωνο Τώρα είσαστε εντάξει, τώρα εντάξει. Λοιπόν, έλεγα ευχαριστώ πολύ σε όλους τους παρόντες, σε όλους τους ομιλητές και σε όλους τους σκιώδεις εισηγητές και συναδέρφους εδώ που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Σημειώσαμε πάρα πολλές σημαντικές ιδέες που θα μας χρησιμεύσουν προκειμένου να βελτιώσουμε τελικά το κείμενο όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας. Υπάρχουν διαφορετικά είδη θυμάτων. Το ακούσαμε αυτό. Έχω μιλήσει με τη συντονίστρια για ε, την εμπορία ανθρώπων, έχω για την καταπολέμησή της δηλαδή, για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής ε, βίας. Όλα αυτά τα θύματα είναι πολύ σημαντικά για μας. Άκουσα γλώσσα πολύ σημαντική για μένα. Ακούσαμε ότι δεν υπάρχει αρκετή δικαιοσύνη, ότι υπάρχει ατιμορρησία μερικές φορές, ότι δεν γίνονται καταγγελίες. Μιλήσαμε για συντονισμό μεταξύ των χωρών ε, μελών ή συντονισμό στο ίδιο το κράτος, ότι τα πράγματα δεν πρέπει να μένουν στα χέρια των οργανώσεων, των εθελοντών. Αυτό λέμε και στη δικιά μου τη χώρα, ότι η ευθύνη είναι του κράτους. Ακούσαμε ότι υπάρχει και ανάγκη για ένα σημείο επαφής. Ενιαίο σημείο επαφής. Και εμείς το έχουμε συμπεριλάβει αυτό στο κείμενο και στις τροπολογίες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας για τα θύματα, λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σημείο επαφής που συντονίζει τη βοήθεια αυτή. Ο συντονισμός είναι πολύ σημαντικός. Ακούσαμε και για την εναρμόνιση της στήριξης, γιατί ανάλογα με το σε ποια χώρα σε περιφέρεια βρίσκεται κανείς, στηρίζεται διαφορετικά ως θύμα. Και σχετικά με την εναρμόνιση, ακούσαμε και για ένα ταμείο, ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα ταμείο για τα θύματα της τρομοκρατίας. Να μην υπάρχει αυτός ο εφιάλτης στον οποίο αναφέρονται τα θύματα, τα οποία γίνονται δεύτερη και τρίτη φορά θύματα και στιγματίζονται μάλιστα. Και μάλιστα αυτό το στιγματισμό εγώ το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Και τώρα, η κυρία Στίβενς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα είμαι σύντομη. Θέλω να ευχαριστήσω εγκάρδια την κυρία που μίλησε για το θάρρος της να έρθει εδώ και να μας μεταφέρει τις εμπειρίες της. Είναι φοβερά αυτά που ζήσατε και οι ελλείψεις με τις οποίες ήρθατε αντιμέτωποι. Στο Βέλγιο είμαστε εννοείται και η κοινωνία και το κράτος έχουν την υποχρέωση να στηρίξουν και να βοηθήσουν κάτι το οποίο δεν έγινε από ό,τι φαίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει η βοήθεια να είναι απευθείας, αμέσως, ξεκάθαρη. Πρέπει να βοηθούμε απευθεία στους ανθρώπους που έχουν περάσει αυτά που περάσατε εσείς. Δεν πρέπει τα θύματα να νιώθουν ε, ενοχές για αυτό το οποίο ζουν. Είναι απαράδεκτος ο τρόπος με τον οποίο σας αντιμετώπισαν. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες μέλη να εφαρμόσουν όσο γίνεται καλύτερα την οδηγία αυτή. Παντού στην Ευρώπη ανεξάρτητα από το που βρίσκεται κανείς, πρέπει να χαίρει της ίδιας στήριξης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάντως που ήρθατε και μιλήσατε έτσι ανοιχτά για την εμπειρία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις. Έξι λεπτά μας απομένουν. Η ε, κυρία Βασιλιάδου δέχτηκε άμεσο ερώτημα και η κυρία Κράχουλετς. Τρία λεπτά η καθεμία λοιπόν έχετε. Κυρία Βασιλιάδου, Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την ερώτηση. Πράγματι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η οδηγία αφορά ελάχιστα πρότυπα, έξοχο εργαλείο παρόλα αυτά. Είναι ένα εργαλείο όπου ποικίλει η εφαρμογή από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Αυτό που κάνουμε μέσω της ανακοινώσεως που δημοσιεύσαμε στις 4 Δεκεμβρίου σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι προσπαθούμε πράγματι να βρούμε τρόπους υποστηρίξεως των κρατών μελών στο έργο που πρέπει να επιτελεστεί. Πράγματος χάρη, θα θέλαμε να μπορούμε να υποστηρίξουμε ε, μέσω κατευθύνσεων προς τα κράτη-μέλη και πιο συγκεκριμά για έμφυλα μέτρα για την υποστήριξη των θυμάτων. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιδών Δικαιωμάτων να δώσουμε προσανατολισμούς για να βελτιώσουμε τη συνεργασία με στόχο να αποφευχθεί το εμπόριο παιδιών. Θα αναθεωρήσουμε το πώς λειτουργούν τα εθνικοί μηχανισμοί παραπομπής και αναπομπή σε διεθνές ε, και εθνικό επίπεδο για να μπορούν να εντοπίζονται τα θύματα. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να προωθούν αρχές που αφορούν το εμπόριο ε, των ανθρώπων, να κινηθούν σωστά επιχειρησιακά, δώσουμε χρήματα για δημιουργία δυνατοτήτων και ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Θα πρέπει τελικά να βασιστούμε από αυτόν. Λοιπόν, ε, όπως λέμε και στην έκθεση υπερενσωματώσεως στην ε, στην ομοθεσία κρατών μελών, μέσω κατευθυντήριων γραμμών, μέσω συμβουλών. Θέλουμε να προωθήσουμε τα παρατεθέντα μέτρα, θέλουμε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη καλύτερη εφαρμογή των μέτρων. Αυτό βέβαια είναι στο επίκεντρο των εργασιών που πρέπει να γίνουν και γι' αυτό δημοσιεύθηκε αυτή η ανακοίνωση. Θα σταματήσω λοιπόν στο 1,5 λεπτό και ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Κράχουλεξ έχει το λόγο. Θα απαντήσω για το θέμα το ψυχολογικό αν είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Όπως είπα, μετά που έφυγα από το νοσοκομείο στην Αμβέρσα, δεν πήρα καμία συμβουλή σε πώς να βρω ψυχολόγο σε μια ξένη χώρα που να είναι ειδικό στις μετατραυματικές αντιμετωπίσεις. Οι συνάδελφοί μου ε, με βοήθησαν να βρω ένα δίκτυο αγγλόφωνο και οι φίλοι μου στις Βρυξέλλες με βοήθησαν. Αναμφισβήτητα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πιο σημαντικό είναι και από πλευράς πρακτικής. Πώς να βρει κανείς τους πραγματικούς ειδικού. Επέστρεψα στην εργασία μου το 2016 τον Οκτώβριο με μερική απασχόληση και θα πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είχα ανακάμψει πλήρως και εργάστηκα με μερική απασχόληση. Θεωρούσα ε, τη δουλειά μου σαν τη μισή μου ανάκαμψη. Μπορούσα να εστιάσω εκεί την προσοχή μου και αυτό βοήθησε και την κόρη μου, διότι περίμενε να επιστρέψει στην πραγματικότητα η κόρη μου και βρήκα ότι ήταν χρήσιμο να επιστρέψω στην εργασία μου. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονες, ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Μας δώσατε πολύ τροφή προσκέψη λόγω της έρευνας που κάνατε και λόγω των προσωπικών εμπειριών περιγράψατε. Πολύτιμα στοιχεία για τα μέλη της Επιτροπής μας. Και εγώ, λέει η κυρία Μπλισκεβισκιούτε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν, όσους πήραν το λόγο, όλα τα μέλη, τους συνεισηγητές, τον συμπρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτή η ακρόαση είναι σημαντικότατη για τους συνεισηγητές και βοηθά να προετοιμάσουμε μια πολύ καλή έκθεση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ πολύ.